Hello, hello dear colleagues. Γεια σας αγαπητοί συναδέλφοι, καλώς ορίσατε στην σημερινή μας συνεδρίαση. Λέει ο Πρόεδρος. Όχι, όχι αυτό. der Entwurf der Tagesordnung ist Ihnen zugegangen. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη. Τη προηγούμενη εβδομάδα τη συνεδρίασης μας έχει μείνει η αντιπροσωπεία στην ΑΕΤ. Θα ήθελα να το κοιτάξουμε στο σημείο 3. Γιατί μάλλον κάποιοι συνάδελφοι έχουν καθυστερήσει στην κίνηση για την ψηφοφορία. Για την ημερήσια διάταξη καταρχάς λοιπόν, να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε. Να ακολουθήσουμε αυτά που συμφωνήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και να ψηφίσουμε, να συζητήσουμε το θέμα που μας έμεινε από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, άρα και αποφασίζεται αυτή η αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Για τις ε, γλώσσες που διατίθενται, να σας ε, πω ότι πέρα από τις γλώσσες που διατίθενται, η συνεδρία μεταδίδεται και στο διαδίκτυο. Και μετά από τις ψηφοφορίες να σας υπενθυμίσω ότι θα γίνουν και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Να σας ζητήσω λοιπόν να κοιτάξετε αν έχετε την ηλεκτρονική σας κάρτα για τις ψηφοφορίες. Και περνάμε έτσι στο 3, στο 3α. Έχετε μπροστά σας ε, τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 9ης Φεβρουαρίου 2012 και τα πρακτικά της 28ης-29ης Φεβρουαρίου του 2012. Όλα αυτά τα λάβατε μέσω email στις 23 του. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, ενστάσεις για τα πρακτικά αυτά, θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν έτσι στο 3α. Η Επιτροπή για τον Έλεγχο Προπολογισμού απέστειλε την προσωπία στην ΑΕΤ για έλεγχο της δαπάνης των ευρωπαϊκών πόρων 22 έως 26 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε αυτή η επίσκεψη και σκοπός βασικά ήταν να διαπιστωθεί ότι τα μέσα τα οποία διατέθηκαν στην ΑΕΤ μετά το σεισμό χρησιμοποιήθηκαν καταλήλως. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση, θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι σημαντικό και καλό θα είναι να το εξηγήσουμε στο σημείο αυτό, ότι τέτοιες διερευνητικές ε, αποστολές είναι ενημερωτική φύσεως και είναι απαραίτητες για το Κοινοβούλιο προκειμένου να σχηματίσουμε μια εικόνα για το τι επικρατεί επί τόπου σε ό,τι αφορά για τις, τις δημόσιες προμήθειες, την δαπάνη των δημοσίων χρημάτων και θα ήθελα να ευχαριστήσω ως πρόεδρος της Επιτροπής τα μέλη της αντιπροσωπείας που έκαναν ένα ταξίδι τέτοιο με διήμερη μόνο παραμονή σε μια τέτοια δύσκολη χώρα. Ξέρετε δεν είναι διασκέταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πολλές οι δυσκολίες που πρέπει να υπερβληθούν σε τέτοιο κλίμα. Θα ευχαριστήσω λοιπόν και τη γραμματεία αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν. και την κυρία Γκέμπορ Γκρέσλε, ιδιαίτερος, που ήταν ε, υπεύθυνη για την αποστολή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσει για το θέμα αυτό, για την επίσκεψη στην ΑΕΤ. Η κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ, πρόεδρε. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για πρώτη φορά ασχολήθηκε με τα μέσα ΕΚΟ. Γιατί σε περίπτωση ανθρωπιστικής βοήθεια ασφαλώς ε, είμαστε λίγο στα όρια και δεν πίστευα να σας πω την αλήθεια ότι το ταξίδι θα ήταν τόσο ενδιαφέρον όσο τελικά μας φάνηκε. Χάρηκα που καταβάλαμε την προσπάθεια, ήταν μεγάλη προσπάθεια για να ταξιδέψουμε εκεί και είδαμε εξ αρχής ότι η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ε, μια βοήθεια που μας δίνει ευγνωμοσύνη, που μάλλον ε, ε αναγνωρίζεται με ευγνωμοσύνη και που δεν αναγνωρίζεται με ευγνωμοσύνη, γιατί ισχύει δύο-τρία χρόνια, αλλά ο κόσμος μας είπε, για παράδειγμα, σε πρώτη φάση ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα. Οι τοπικές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις μας το είπαν αυτό εξ αρχής. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Κοιτάξτε, διακόπτη κυρία Γκρέσλα, μήπως θα μπορούσατε να πάτε λίγο παραπέρα για να μιλήσετε. Ναι, αν θα θέλετε παρακαλώ να μετακινηθείτε λίγο ή να σιωπήσετε. Συνεχίζει η κυρία Γκρέσλε. Η ΑΕΤ είναι μια χώρα η οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, στην οποία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση. Ο σεισμός ε, βελτίωσε κάπως ε, την κατάσταση γιατί ενώ πριν τον σεισμό είχε πρόσβαση σε γιατρούς μόνο το 30% τώρα είναι 60% από ανθρωπιστικής απόψης δηλαδή, ε, βρισκόμαστε σε μία παγίδα. Με κάθε μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας και μετά από δύο χρόνια αναγκαστικά πρέπει να μειώσουμε τα ποσά. Με κάθε μείωση λοιπόν ε, διατρέχουμε τον κίνδυνο στην προηγούμενη κατάσταση. Και αυτό το συνειδητοποιούμε, το αντιλαμβανόμαστε. Και είδαμε ότι αν δεν βελτιωθεί η πολιτική κατάσταση στην IT δεν πρόκειται ε, όση βοήθεια και αρρωγή και να χορηγηθεί να καταφέρουμε να αλλάξουμε κάτι με μόνιμο τρόπο. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με μία μόνιμη διαρκή αλλαγή της κατάστασης. Αυτά είναι τα δύο ενδιαφέροντα σε μία για το πώς θα συνεχίσουμε δηλαδή σε τέτοια θέματα. Πώς θα συνεχίσουμε σε ό,τι αφορά την, ανθρω... την ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα αυτή. Συναντηθήκαμε με όλου του σημαντικού παράγοντε επιτόπου και είδαμε ότι η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί απεβίωσε κατά το σεισμό η διευθύντρια και υπήρξε μία αλλαγή στην ηγεσία. Έχουμε κάποιον ο οποίος θα εκπροσωπήσει την ε, πρέσβη μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε τρία άτομα τα οποία αλλάζουν στην ηγεσία της ε, αντιπροσωπείας. Αυτό δεν είναι θετικό και θα πρέπει να το σκεφτούμε. Συναντήσαμε υπαλλήλου πάρα πολύ δεσμευμένου και οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν με θαυμαστό τρόπο για τη χώρα, αλλά είδαμε επίσης ότι είναι απολύτως απαραίτητο και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ε, εργασίας της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου. Γιατί οι μεγάλοι δωρητές έχουν παρατηθεί ουσιαστικά από την δεκαετία των 90 από την IT. Και αυτό πρόκειται, εδώ πρόκειται για ένα σημείο το οποίο δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε, γιατί χωρίς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προκειμένου να βελτιωθούν, να ενισχυθούν οι τοπικές δομές, προκειμένου ο κόσμος να λάβει πολύ περισσότερες ευθύνες από ό,τι ως τώρα. Εγώ προσωπικά και είναι η προσωπική μου άποψη αυτή, πάντα είχα ένα δυσίωνο συνέστημα αν θέλετε σε περίπτωση αποδυνάμωσης του τοπικού πληθυσμού. Αμφιβάλλω πάρα πολύ για το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η σύστασή μας λοιπόν, οι συστάσεις μας είναι σαφέστατες. Συστήνουμε να ενισχυθούν οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αυτοδιοίκησεις, οι τοπικοί φορείς, να μην αναγκάσουμε τις κυβερνήσεις της αυτοδιοίκησης να συνεχίσουν με τον τρόπο που λειτουργούν ως τώρα. Ακούσαμε από την Παγκόσμια Τράπεζα ότι η κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει ένα υπολογιστικό σύστημα μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ανιχνευσιμότητα των πόρων από τους, και πώς δαπανώνται από τις δημόσιες αρχές. Όλα αυτά, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά και διακυβεύουν ε, τις παγκόσμιες χορηγήσεις από τους δωρητές. Υπάρχει επίσης ε, έντονη επιθυμία να αναλευτούν ευθύνε ε, υπό τον όρο φυσικά ότι πληρούνται οι σχετικές ε, οι σχετικοί οι σχετικές συνθήκες. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στην ΑΕΤ. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία, να χρησιμοποιήσουμε την τρέχουσα κατάσταση. Και συμφωνήσαμε και στα συμπεράσματα, μάλλον ε, ένα συμπέρασμα δεν μας βρήκε απόλυτα σύμφωνο, στο τρίτο, όπου αναφέρεται ότι αν ε, δεν πληρεί η κυβέρνηση τους όρους αυτούς, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την βοήθειά μας. Ε, κάποιοι συνάδελφοι δεν συμφώνησαν, αλλά από την άλλη, αν δεν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, κάτι θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Νομίζω ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η επίσκεψη, ότι ήταν σημαντικό τα χρήματα να δαπανηθούν, να επενδυθούν στην βοήθεια των σεισμόπληκτων για, ε, το νερό, για τις εγκαταστάσεις υγιεινής και ότι Πλέον η IT θα πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο, να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες η ίδια η χώρα. Ξέρουμε ότι χρειάζεται πολλά χρήματα για την ανοικοδόμηση, ότι πολλά πράγματα ακόμα απομένουν να γίνουν και ότι σε θέματα πρόληψης φυσικών καταστροφών και σεισμών ε, δεν έχει γίνει ακόμα καμία πρόοδος και εξακολουθούν να γίνονται τα ίδια σφάλματα που παρουσιάζονταν και πριν. Δηλαδή, ο επόμενο σεισμό θα έχει ακριβώ τα ίδια αποτελέσματα όπω και ο προηγούμενο. Και δεν γίνεται τίποτα ούτε από, τις, ε, από την κυβέρνηση. Είδαμε κάποια σημεία θετικά που μας κάνουν να ελπίζουμε, αλλά από την άλλη πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στην ΑΕΤ. Δεδομένου και το γεγονότος ότι μπλέκουμε σε ένα φαύλο κύκλο των ίδιων σφαλμάτων που θα έχουν τα ίδια αποτελέσματα στην επόμενη φυσική καταστροφή. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα εξακριβώσουμε. Ήταλος δεν είναι βιώσιμη η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, να ευχαριστήσουμε την υπεύθυνη της αντιπροσωπείας. Δεν ξέρω αν θα έκανε ένας άλλος το λόγο. Nur eine, ein, ein Ένα μικρό σχόλιο για αυτά που διαπιστώσαμε. Τα συνοψίσατε ήταν πολύ ακριβή τρόπο. Στη σύσταση 3 έχουμε την εξή διαφορά. Αν παγώσουμε, αν ήταν να παγώσουμε τα ποσά που θα χορηγούνται, δεν θα είχα αντίρρηση. Αλλά η αρχική πρόταση ήταν να επιστραφούν τα χρήματα αυτά. Σύμφωνοι ότι για την χορήγηση και την ε, περαιτέρω μάλλον χορήγηση χρημάτων θα πρέπει να πληρούνται οι όροι που θέλουμε. Ιδάλλως θα παγώσουν τα ποσά αυτά που χορηγούνται. Σύμφωνοι. Αλλά στην κατάσταση που ζει ο κόσμος ακόμα στη χώρα αυτή και είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση, ακόμα και για δύο μέρε που μεταβήκαμε. Και μάλιστα υπό πολύ πλεονεκτικού όρου, Ήταν πραγματικά τραγική η κατάσταση. Δεν μπορούμε να τους απειλήσουμε με επιστροφή των χρημάτων. Νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό, η βασική μας διαφορά. Ευχαριστώ, κύριε Λιμπεράτσκι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά υπόψη τόσο επανήκρες λογικά και επίσης αν κατάλαβα πάρα καλά ε, η κατάσταση πιέζει πάρα πολύ γιατί υπάρχει πρόβλημα ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες ε, υγείας και αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια ε, από, από, από ανθρωπιά. Και τι γίνεται, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει, δεν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι να βοηθούν σε καθημερινή βάση. Τώρα, Εάν κατάλαβα καλά, εάν σταματήσουμε να τους βοηθούμε, τότε θα πεθάνει ο κόσμος, θα πεθάνουν άνθρωποι. Επίσης έχω άλλη μια ερώτηση. Οι, οι άνθρωποι στην ΑΕΤ γνωρίζουν ότι βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Μήπως ξέχασα κάποιον. Όχι. Ωραία λοιπόν, άρα μπορούμε να κλείσουμε. Α, συγγνώμη, μια απάντηση θέλετε να δώσετε. Κυρία Κρέσλε. Α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας απαντήσει από δική της πλευρά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι η διευθύντρια της υπηρεσίας αυτής και φαίνεται πάρα πολύ καλό εάν κάποιοι τελικά ελκύσουν την προσοχή στην χώρα. Γιατί μην έχουμε μόνο αρνητική δημοσιότητα. Και αν κανεί πάει και κάνει αυτό το οποίο έκανα και εγώ τόσα χρόνια από διαφορετικές θέσεις τότε κανείς δεν θα εξεπλήσει το ποιο έκανε αυτό. Αν δηλαδή αυτό το οποίο είδα εγώ, Εάν επίσης ε, ταξίδευε πάνω κάτω την Αφρική όπως εγώ και αυτό το οποίο εντυπωσιάζει είναι όταν κανείς έτσι ενεργεί ε, να αναλάβει την ευθύνη να πάει στην Αιτία και μάλιστα περνώντας τα σύνορα από Δομινικανή Δημοκρατία είναι σαν να γυρίζει πίσω στον χρόνο, να πηγαίνει στον Μεσαίωνα. Έχω πάει στη χώρα. Πήγα αμέσως μετά από εσά. Και για πρώτη φορά είχα την ευκαιρία μετά από τόσα χρόνια να μιλήσω σε έναν υπουργό. Είμαι στον κύριο Μπελερίφα την πρώτη φορά. Δεν μπορούσε να μιλήσει την πρώτη φορά που προσπάθησα να τον βρω και πριν μερικές εβδομάδες λοιπόν μίλησα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Για μένα αυτό είναι ένα πρώτο θετικό σημάδι. Και αυτό το οποίο με ρώτησαν είναι ακριβώς αυτό που εσείς ακριβώς και ρωτάτε. Τι κάνουμε εκεί. Επί δύο χρόνια δρούμε, έχουμε δώσει μια σειρά υποσχέσεων, είμαστε ένας από τους βασικούς δωρητές της Ευρωπαϊκή Ένωση και ο κύριος Λεβεράτσκι είπε είμαστε οι μόνοι δωρητές, όχι, είμαστε οι μόνοι ούτε οι βασικοί γιατί εγώ ήρθα σε επαφή με όλους τους δωρητές. Αν μιλήσετε στους Αμερικανούς, για εκείνους η Αιτή είναι το ίδιο όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Για αυτούς είναι η χώρα κλειδί από πλευράς χώρας που έχουν στοχεύσει για να την βοηθήσουν. Οι Καναδοί επίσης θεωρούν ότι είναι ένα πρόβλημα στο, στον κήπο τους, στο στη γειτονιά τους και θέλουν βοηθήσουν. Γαλλία, Ισπανία. Έχουμε έρθει σε επαφή με όλους αυτούς και όλοι επομένω ξέρουμε τι άλλες προσπάθειες καταβάλλονται, γίνονται εντατικές ε, διαβουλεύσεις. Είναι μια χώρα η οποία ό,τι πρόβλημα υπάρχει τυχόν εκεί γιγαντώνεται. Εκεί η πρόκληση, ο πύχη ούτω η πίνη τη πρόκληση που γίνεται ουδή κανεί είναι πάρα πολύ ψηλά και γι' αυτό και μα πήρε πάρα πολύ χρόνο τόσο ώστε να ξεκινήσουμε τι προσπαθίε μα. Δεν υπάρχει τίποτα που να βρίσκει αντίθετη στο κείμενό σα για του μη κυβερνητικού οργανισμού, για του συμβιβασμού. Δουλεύουμε επομένω με αυτού και τελικά ε, θέσει είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβάλλετε τις προσπαθίες σας. Πάρα πολύ ευχάριστο να είναι εκεί κάποιο και να υπάρχουν εδώ διάφορα σύμβολα να προβάλλετε. Δηλαδή, πολύ σημαντικό είναι αυτό που, που λέμε όριμο φρούτο. Και όταν κανείς δουλεύει εκεί, όμως τελικά προβάλλεται πολύ λιγότερο στην πραγματικότητα. Και ο Επίτροπος Πίμπαλτς, ο οποίος επίσης ε, έχει αναλάβει και σημαίνει κάποια πρόοδο, πήγε την τελευταία φορά στη χώρα, ήταν πρόκειτο για το πρόσφατο ταξίδι. Και... <laughs> Κι όμως, οι υπουργοί στη θέση τους παρόλα αυτά. Και όλοι είπαν ότι θα αφιερώσουν μία ολόκληρη μέρα για να μιλήσουν, για να ανταλλάξουν απόψεις με τον Επίτροπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη απόδειξη Τη προβολή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλή κάτι, κάτι, κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο πέτυχε ο Επίτροπο. Και για μα αυτό είναι η απάντηση στο, στο ερώτημα που θέσατε. Και όταν ξανάρχισα, ε, μίλησα με τον ε, Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών και μου είπαν ε, εσείς, Αμερικανοί, τι κάνετε με τις μη, μη κυβερνικές οργανώσεις, μήπως υπονομεύετε την προσπάθεια και την κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσουμε τα πράγματα γιατί έχουμε κάποιους που όντω έχουν χολέρα, πρέπει να αντιμετωπίσουν. Πρέπει κάποιοι άλλοι να σωθούν από το θάνατο. Με τους αδέλφους της ΕΚΟ λοιπόν κάνουμε ό,τι μπορούμε και λόγω των νευροσπαθικών προσπαθειών <clears throat> κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη χολέρα και επί τόπου. Γιατί είμαστε εκεί και γιατί ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Ο κόσμος που μπορεί να έρθει και να πάρει τα φάρμακα. Και να σα πω έτσι ένα παράδειγμα, εάν παράσχεται. Ελεύθερα ε, δωρεάν υπηρεσίες. Πώς θα πιέσετε την κυβέρνηση. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι μη και μεγιστονώσει δίνουν κάποια λίγα χρήματα και αυτό το οποίο κυρίως μας ε, εντυπωσιάζει είναι ότι πρόκειται για κάποιες συστάσεις οι οποίες και σήμερα ακούστηκαν όσον αφορά το πάγωμα των ε, εκταμείωσεων. Πάρα πολύ δύσκολο να πει η κυβέρνηση να αναγκαστεί να κάνει κάτι, γιατί σε αυτή την περίπτωση τότε η κυβέρνηση θα συμφωνήσει, έτσι για να συμφωνήσει, και κατόπιν θα αθετήσει αυτά τα οποία αποσχέθηκε. Είναι το θέμα εδώ πέρα των ευρωπαϊκών αξιών, είναι θέμα της δέσμευσης, της υπόσχεσης ότι θα πρέπει να την τηρήσουμε και θα πρέπει τις διαδικασίες της να τις ε, βοηθήσουμε. Ας πω ένα σημείο παράδειγμα. Εμείς ξέψαμε τόσα χρήματα όσον αφορά την, ε, ε, στο σχεδιασμό, την, κατασκευή ρόδων. Είδατε εκεί πόσο δύσκολο είναι στο Πόρτο Πρένς και κυρίως εκτός της πρωτεγούσης. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έχουμε σημαίες στο δρόμο. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε σημαίε γιατί οι δρόμοι δεν συντηρούνται σωστά. Οπότε τους κάνουν τα λάστιχα και λένε «Α, αυτοί οι παλιοευρωπαίοι χτίσαν αυτούς τους παλιοδρόμους». Άρα τι κάναμε. Διαπραγματευθήκαμε με τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης και προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα ενεργοποιηθούν τα χρήματα αυτά για την συντήρηση των δρόμων. Άρα θα πρέπει κανείς να περάσει από το κοινοβούλιο, θα πρέπει να επιφέρει κάποιε αλλαγέ, να γίνουν οι σχεδία ψηφοφορίες, κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο. Όπως είπαμε για πρώτη φορά, για πρώτη φορά που εγώ πάω εκεί βρήκα κάποιον να μιλήσω, είχα συνομιλητέ. Και για πρώτη φορά επομένω στήσαμε, συγκροτήσαμε αυτό το Ταμείο Συντήρηση των Δρόμων. Άρα υπάρχουν αλλαγέ προ το καλύτερο που μπορείτε να δείτε. Εμείς αυτά τα κάνουμε μέσω της υποστήριξης από τον προπολογισμό, γιατί αλλιώς το Κοινοβούλιο θα έχει τα χέρια σταυρωμένα αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Και μιλούμε για κάποιες ε, μικρές υπηρεσίες, οι οποίες και αυτές θα ε, σταματήσουν. Οι Ιαπωνέζοι, Νορβηγοί και αυτοί εισφέρουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός δωρητής. Δεν είμαστε όμως οι μόνοι. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η χώρα αρχίζει να υλοποιεί κάποιες δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις. Είναι μεγάλο το δήμα που έγινε. Η χώρα δεν είναι τη μάχη της. Λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις μας, τις σκληρές συστάσεις, αλλά έχουν την πρόθεση να τα υλοποιήσουν όλα αυτά. Πρόκειται για τα πρώτα βήματα όσον αφορά κάποια μέτρα εισοδηματικής πολιτικής. Κάτι έχουμε κάνει. Θεωρούμε ότι πάμε καλά. Είπατε κάτι για την ετοιμότητα όσον αφορά τις θεομηνίες, τις φυσικές καταστροφές. Γιατί, όπως ξέρετε, ε, είναι ε, τρομερές οι καταστροφές που έχουν χτυπήσει τη χώρα. Έτσι λοιπόν κάποιοι θα πρέπει να πάνε σε αυτή την ε, όμορφη χώρα Μιλούμε για κάποια 15 εκατομμύρια που διατέθηκαν μέσω του χρηματοδοτικού μέσου, τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πολιτική προστασία, να υπάρχει ετοιμότητα για να αντιδράσει κανείς όσον αφορά τις θεομηνίες. Επίσης, αναφέρεται τα προβλήματα της στέγασης. Φερρυπίν, ε, έχουμε για το Γεωστατικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Έχουμε ένα σωρό υπέροχα όργανα που τους δώσαμε, τους εκπαιδεύσαμε, το, αυτό το, αυτή τη δημόσια υπηρεσία της γεωστατικής. Όμως έγινε σεισμός. Μετά το σεισμό δεν έμεινε τίποτα. Ούτε κτίριο, ούτε προσωπικό, ούτε τα όργανα τα οποία τους εδωρήσαμε. Ανασυγκρότηση έχει αρχίσει, ανοικοδόμηση έχει αρχίσει σε νέες αρχές, σε νέες βάσεις επικεφαλής είναι ο ΟΗΕ, η ανερμόδια υπηρεσία που έχει βοηθήσει πάρα πολλές χώρες που έχουν πληγεί από το σεισμό και όλοι οι δωρητές συνεφώνησαν με αυτή την προσέγγιση. Και επομένως έχουμε εδώ συγκεκριμένη παράδοση για το πώς θα ξαναχτιστεί το πρώτο Πρένς. Άρα αντιδρούμε σε αυτές τις προκλήσεις. Δεν πρόκειται για ένα παγκόσμιο, ένα σφαιρικό υδατοστεγές, ας το πούμε, αλάθη το σχέδιο. Όμως προχωρούμε όσον αφορά τον χώρο ταξικό σχεδιασμό. Δεν είναι εύκολο, τίποτα δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω γιατί έχουμε πολλά θέματα. Α, καλά, καλά. Πάντως, ήμασταν εκεί. Θα είμαστε εκεί. Δεν είναι εύκολο. Μας επικρίνουν. Δεν υπάρχει μόνο ευγνωμοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι η τηλεόραση έχει πάψει να προβάλλει το πρόβλημα και ο κόσμο, τι είναι να ξεχάσει μέχρι ότου έρθει η επόμενη ανθρωπιστική καταστροφή. Εμεί είμαστε εκεί, θα πρέπει να εργαστούμε με την κυβέρνηση, αλλιώ όπω ο ίδιο αναφέρεται δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι η χώρα πιο έτοιμη ούτω ώστε να αντιμετωπίσει τι φυσικέ καταστροφέ. Είδαμε τι έγινε με το Σαν Σαλβαδόρ, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τη χώρα να ετοιμαστεί για αυτό τη φυσική καταστροφή και μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στην Αιτία. Επιτρέψτε μου άλλα δύο θέματα να θίξω. Πρώτα-πρώτα αυτό το οποίο εσείς ζητήσατε για αναθεώρηση του προγράμματος και κατά την επίσκεψή μου είδαμε ότι έχουν χαθεί αρχεία. Ξαφνικά ξαναβρέθηκαν. Εμείς για να δούμε τι πριν από 15 χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχουν καταστραφεί πάρα πολλά αρχεία. Επίσης έχουμε άλλους κανόνες ε, με την απαλλαγή όσον αφορά τον χρηματοοικονομικό έλεγχο. Θα έπρεπε να μην έχουν χαθεί τα έγγραφα Πρόκειται για συσήφιο έργο και μέχρι ένα σημείο θα, θα το καταφέρουμε να δούμε όμως. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε που να είναι και αξιόπιστο επί τη βάση των προτεραιοτήτων που έχουμε τάξει για τη χώρα. Κάτι άλλο τώρα πρέπει να σας αναφέρω. Όταν άρχισαμε να δουλεύουμε, διαπιστώσαμε η ΕΚΟ πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Και πρόκειται για δύο επιτρόπους, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί και είπαν, ο Πίτρος α πούμε, Ας προσπαθήσουμε, ας ε, διασυνδέσουμε την ΕΚΟ με την ανάπτυξη και να δώσουμε προτεραιότητα στην IT. Αν μιλήσετε επί τόπου στον κόσμο θα καταλάβετε ότι αυτά που έχουμε πετύχει δεν τα έχουμε καταφέρει πουθενά Και οι περιορισμοί υπάρχουν σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε στη χώρα και γενικά τι μπορούμε να κάνουμε με τα μέσα πολιτική μας αν γίνεται να ξαναδούμε τις ε, συστάσεις, όπως είπατε και εσείς, ότι λέει η έκθεση άγγιξε τις πιο ευαίσθητες χορδές όλων όσων νοιάζουν τη χώρα αυτή. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Μπουτικεβιτσκένα. Για την έκθεση αυτή η ε, παρουσιάστηκα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και είναι σαφής ότι το έργο σας ε, εκεί είναι πολύ δύσκολο. Κλείνοντας τώρα, θα ήθελα να δώσω το λόγο εκ νέου στην κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση που, αποτελούν, που αποτελεί ένα μικρό παράδειγμα των όσων ζήσαμε και εμείς εκεί. Ζήσαμε και είδαμε ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες είναι πολύ σε πολύ άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ καλή περιγραφή της κατάστασης. Έτσι έχουν τα πράγματα πράγματι. Η κριτική μας δεν είναι κριτική σε αυτά που πραγματοποιούνται επί τόπου, όχι. Η αποτελεί μια απόπειρα να εξηγήσουμε το τι θα πρέπει να γίνει και τι θα πρέπει να προσέξουμε τον επόμενο καιρό. Γιατί είδαμε ότι με όλη την καλή θέληση που υπάρχει, γιατί υπάρχει, αν και εξαρτάται από τον κάθε φορέα, πέρα από την καλή θέληση λοιπόν θα πρέπει να ε, υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα και από την κυβέρνηση. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτή την κριτική μετά από αυτά που ζήσαμε. Αν και αναρωτιέμαι μήπως αυτή η προσωπική κριτική είναι κάπως υπερβολική. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλοι ήμασταν ευγνώμονε για όλα όσα γίνονται εκεί υπό δύσκολε συνθήκε και ότι θέλουμε να τονίσουμε ότι για το μέλλον υπάρχουν ασφαλώς ε, κάποιες προκλήσεις και θα πρέπει να μάθουμε από τα παθήματα του παρελθόντος και ίσως στις μελλοντικέ προκλήσεις θα πρέπει να αντιδράσουμε με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ως τώρα. Συνδεθήκαμε με την επιστροφή μας με τον Επίτροπο Πίπαλξ και με την, κυρία, με την Επίτροπο Γεωργίβα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι βέβαιη ότι πάντα θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα αυτό και ότι σίγουρα δεν πρέπει να ξεχάσουμε την ΑΕΤΗ. Ήταν υπερβολικά έντονα αυτά που ζήσαμε για να τα ξεχάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Αποδεικνύεται ότι και στον τομέα αυτό είναι σημαντικό να τοποθετούμαστε ως Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Πρόκειται για αξιολόγηση. Μάλλον εκτιμούμε την ε, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρώ ότι ο ρόλος μας είναι σωστός και είναι προς το συμφέρον των φορολογούμενων και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το μεταφέρουμε προς τον πολίτη, ότι κοιτάξτε θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι δαπανώνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρήματα του φορολογούμενου προ όφελο όλων όσων μα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και να περάσουμε σε ένα μεγάλο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ψηφοφορίε. Θα μα απασχολήσει αυτό το θέμα αρκετή ώρα. Μεγάλο μέρος των ψηφοφοριών θα γίνουν ηλεκτρονικά για να έχουμε και σαφή αποτελέσματα. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία αν θέλετε. Δοκιμαστική λοιπόν ψηφοφορία αν θέλετε. Να κάνουμε ένα τεστ. Έναρξη ψηφοφορίας. Μάλιστα. Πέρας. αλλά φαίνεται να είναι μια χαρά. μέλη έχουμε. Okay. Ja, wir starten mit. Να ξεκινήσουμε με την απαλλαγή. 2010 Gesamthaushaltsplan der EU, Einzelplan 3. Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τμήμα 3, Επιτροπή. Εισηγητή, ο κύριο Χέλνερ. Long, uh, on this, but I Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. Νομίζω ότι πρώτα όμως να πω ότι έχει ε, υπάρξει πάρα πολλή δουλειά για πάρα πολλούς ανθρώπους. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους κοιόδης εισηγητές Νομίζω ότι διασκεδάσαμε σε εισαγωγικά όλοι μαζί, αλλά κάτι πετύχαμε. Θα ήθελα επίσης με αυτή την αφορμή να ευχαριστήσω τον Μπεν, τον Τζόνας, τον Κριστόφ, γιατί νομίζω ότι χωρίς τη βοήθειά τους και την ικανότητά τους δεν θα είχα πετύχει πολλά πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες, ελπίζω πολλές να κερδίσω και λίγες να χάσω, αλλά εν πάση περιπτώσει ανεξαρτήτως της έκβασης των ψηφοφοριών, η έκθεση θα είναι καλή έκθεση. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Το πιο σημαντικό πάντως είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει, είναι το αν θα δώσουμε ή όχι απαλλαγή. Εμείς έχουμε βάλει δύσκολα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπαμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να τα δεχτεί θα δώσουμε την απαλλαγή. Αυτό ε, είχαμε πει. Πήραμε μία επιστολή από τον κύριο Σεμέτα ο οποίος νομίζω απάντησε καλά, ανταποκρίθηκε στα ερωτήματά μας. Σε δύο παραδείγματα να σας δώσω πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Το πρώτο να σας πω το εξής είναι το θέμα της κοινή διαχείρισης και της κοινή ευθύνη. Η μοιρασμένη ευθύνη όμως για μας δεν είναι ευθύνη. Δεν μπορεί να στρέφει το δάκτυλο στα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λέει αυτή είναι η αμαρτωλή και από την άλλη τα κράτη-μέλη να λένε ότι εμείς σκοτιστήκαμε για το αν θα πάρει η Επιτροπή την απαλλαγή. Δεν πάει πουθενά έτσι. Εμείς περιμένουμε να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Έχουμε πολλές ελπίδες για το επόμενο πλαίσιο, ιδιαίτερα για τη Γεωργία και το Περιφερειακό Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό λέει ότι θα κάνει, θα χρησιμοποιήσει τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της. Αυτό λέει ο ΣΕΜΕΤΑ. Βέβαια εμείς είμαστε συνομοθέτες και μας ρίχνει και σε μας ευθύνη ο ΕΜΕΤΑ. Αλλά σε σχέση με το επόμενο νομοθετικό πλαίσιο νομίζω ότι έχουμε κάποιες εγγυήσεις έτσι ώστε να μην ξαναγίνουν πια τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Ε, δεν μπορούμε να λέμε ότι τα ίδια κράτη μονίμως αμαρτάνουν χωρίς να υπάρχει καμία βελτίωση από έτος σε έτος. Λοιπόν, Έχω την εντύπωση ότι αυτά τα οποία συνέβησαν το 2010 δεν ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Είχαμε ελλείψεις στον τομέα της πληροφόρησης, είχαμε ελλείψεις στον τομέα της γνώσης και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναγνωρίζει αυτό. Γι' αυτό χαίρομαι λοιπόν που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρξει προσεκτική εξέταση του τι πήγε άσχημα στο προηγούμενο πλαίσιο χρονικό και να μας δώσει από εδώ και πέρα πολύ περισσότερη και καλύτερη ενημέρωση για τα χρηματοδοτικά μέσα. Γιατί αυτά είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον. Πάντως, επαναλαμβάνω, η απάντηση στη δική μας έκκληση ήταν καλή από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει νομίζω να δώσουμε την απαλλαγή. Να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και τώρα να περάσουμε στις ψηφοφορίες και να πω εξ αρχής το εξής. Ο εισηγητής έχει υποβάλει δύο δυνατότητες, είτε αναβολή, είτε χορήγηση της απαλλαγής. Τα αιτιολόγησε και τα δύο σενάρια. Θεωρεί ότι είναι δικαιολογημένη η χορήγηση απαλλαγής, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει με τη διαδικασία ψηφοφορίας. Η διαδικασία είναι ε, η εξή. Αν ψηφιστούν ε, οι τροπολογίες 1 και 2, θα γίνει αναβολή. Αν δεν αποφασιστεί η αναβολή, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Η σύσταση δεν θα υπάρξει επιπλέον ψηφοφορία γι' αυτό. Έτσι εκτιμώ ως πρόεδρο την κατάσταση. Συμφωνείτε με τη διαδικασία αυτή από τη δικαστική απόψη. Γιατί έχει συνέπειες η απαλλαγή, η αναβολή. Θα σήμαινε τη λήψη του ηλικής απόφασης στο φθινόπωρο. Και αν ε, δεν το αποφασίσουμε αυτό, ουσιαστικά αποφασίσουμε η απαλλαγή. Αν λοιπόν συμφωνείτε να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες 1 και 2 που είναι ταυτόσιμες. Έναρξη ψηφοφορίας. So, die Abstimmung ist geschlossen. απορρίπτεται η τροπολογία. Και άρα απορρίπτεται η αναβολή και ουσιαστικά συστήνεται η χορήγηση απαλλαγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλάζει λοιπόν η απόφαση μέσω της τροπολογίας Όποιο συμφωνεί με το σύνολο του ψηφίσματο, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Α, του αριθμού. Ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Αν ψήφισατε όλοι. Okay. With, uh, okay, I didn't vote. Okay, <laughs> sorry. Um, vote is closed. Ωραία. Δεύτερη πρόταση για την απόφαση να ψηφίσουμε την ε, αναβολή της χορήγησης 5 και 6 έναξη ψηφοφορίας αν ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας ωραία άρα απορρίπτεται και άρα κατά συνήπεια αποφασίζονται και εγκρίνονται οι 7 και 8 τροπολογίε. Έχουμε και τη, τη λογική σκέψη 8 τροπολογία 9 να ψηφίσουμε ωστόσο ηλεκτρονικά για την τροπολογία 9 παρακαλώ. Vote is, vote is open. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας τώρα. Εγκρίνεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία για το σημείο αυτό. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, ένα ψηφοφορία. is closed. Πολύ ωραία. Αν ψήφισατε όλοι, πέρα ψηφοφορία. εγκρίνεται. Στο 3 τώρα. 10 και 11 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες Απερίφθη. Οπότε θεωρείται ότι δίδεται η απαλλαγή και πρέπει να ψηφίσουμε τώρα την 14. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική στην 14. Hat jeder abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Klaus, Abstimmung ist geschlossen. Πέρασε τη ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά, συνολική τελική ψηφοφορία. Jeder abgestimmt. Vote Αν ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφορίας. Okay. Damit Ziffer. Ωραία και πάμε λοιπόν στο 4. 15 και 16 τροπολογίες. Αναβολή. Ψηφίζονται ηλεκτρονικά. Αν ψήφισατε όλοι, πέρα ψηφοφορίας. Ε? Απορρίπτεται. Ναι, Άρα θεωρείται ότι χορηγείται η απαλλαγή. Πάμε στην 19, έναρξη ψηφοφορία ηλεκτρονικά για το 19. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα σύνολο επί του συνόλου της πρότασης απόφασης αποτροποποιήθηκε. Αν ψήφισατε όλοι, πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5. Τροπολογίες 20 και 21. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρα χορηγείται η απαλλαγή. Να ψηφίσουμε την 14, λέει ο Πρόεδρος. Ηλεκτρονικά 24, 24. Ηλεκτρονικά την 24. Αν ψηφίσατε όλοι. Ελλάδα. Πέρα ψηφοφορία. Τώρα το σύνολο της απόφασης, ηλεκτρονικά αν θέλετε, πέρα ψηφοφορία. Αν ψήφισατε όλοι. Α, όχι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 6. 25 και 26. Ταυτός είναι τροπολογίες. Ηλεκτρονικά να ψηφίσουμε έναρξη ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρα θεωρείται ότι χορηγείται η απαλλαγή και περνάμε στην 29 τώρα. Ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Άρα, να ψηφίσουμε την τροποποιημένη απόφαση. Ηλεκτρονικά, έναρξη. Πέρας. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα τώρα εκτελεστική υπηρεσία. Στο 7. Να ψηφίσουμε 30 και 31 ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απορρίπτεται. Mm. Χορηγείται λοιπόν η απαλλαγή. Να ψηφίσουμε το 34 ηλεκτρονικά. Ναι, ναι. τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. Τώρα το σύνολο τη απόφαση όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Πρόταση αποφάσεων 8. 35. Αναβολή. Άρχεται η ψηφοφορία για την 35. Ηλεκτρονική ψήφος. Everybody voted. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 36 και 37 συνεπώς είναι ταυτόσιμες. Θεωρούνται δεκτές. Περνάμε στη 38. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 38. Ψηφίζεται. Πέρας της ψηφοφορίας. Δεκτή. Ψηφίζουμε το σύνολο της τροπολογημένης πρότασης ηλεκτρονική ψήφος. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Πρόταση ψηφίσματος 9 λοιπόν. Τροπολογία 211. Ηλεκτρονική ψήφος. Everybody voted. Vote is closed. Τέλος. Απορρίπτεται. Τώρα να ψηφίσουμε διανάταση του χειρός. Παράγραφος 2, τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43, 44, 45, 46 από κοινού. Εφόσον συμφωνείτε να τις ψηφίσουμε από κοινού. Για μια στιγμή λέει ο πρόεδρος. 43 μέχρι και 45, όχι 46. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 46. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Απορρίπτεται. 47. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι 50, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 51, υπέρ, κατά, αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 51. Electronic vote is closed. Τέλος. Σαφώς γίνεται δεκτή, έκανα λάθος εγώ λέει ο Πρόεδρος. Συμβιβαστική τροπολογία τώρα, ένα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 52 καταπίπτει, περνάμε στην 53. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 54. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή γενικά. Γίνεται δεκτή. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 56 υπέρ. Α, για μια στιγμή, για μια στιγμή. 56 με 59 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα έχει ζητηθεί ξεχωριστή ψηφοφορία σε, δι... σε τρία τμήματα της 60. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα της 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό αλλά μπορεί να υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα. Όχι, δεν πειράζει. Το τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 62, 63 και 64. Ποιοι είναι υπέρ. Όχι, α, υπάρχει διαφωνία. Ξεχωριστά θα τις ψηφίζουμε. 62 πρώτα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 66 παρακαλώ ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. Βιάστηκα λίγο λέει ο Συμβιβαστική τώρα 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Η 67 καταπίπτει. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 68. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Δεκτή. 69. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 74 έχει αποσυρθεί. Α, έχει καλυφθεί μάλλον. Η 75. Υπέρ. Αποχές. Δεκτή. Κατά, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος, τα μπέρδεψα. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι, κατά. Ο πρόεδρος ξεχνάει το κατά. Εβδομήντα έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εβδομήντα επτά. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεν κατάλαβα. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 80. Ψηφίστε. Τέλος. Δεκτή. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 82. Τέλος. Απερίφθη. 83 και 84. Ταυτόσιμες υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. 85 υπέρ κατά, αποχές, δεκτό. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 89 προφορική τροπολογία της Ingeborg Gressler δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Εδώ ξεχωριστή ψηφοφορία στην 90. Πρώτο τμήμα. Προφορική τροπολογία της Μακοβέη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Το δεύτερο τμήμα τώρα της 90. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα. Με την προφορική τροπολογία Μαρινέσκου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 92 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να παίρνετε μέρος στην ψηφοφορία διανατάσεως. Δεν καταλαβαίνω αλλιώς. Ποιοι είναι υπέρ της 92. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 92. Ψηφίζουμε και ελέγχουμε. Τέλος, απερίφθη με μικρή διαφορά. 93. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 94. Υπέρ. Α, για μια στιγμή. Για μια στιγμή διορθώνει ο πρόεδρος. 102. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. από κοινού ψηφιοφορία από 105 μέχρι και 109. Όχι, υπάρχει κάποια διαφωνία. Οπότε θα ψηφίσουμε ξεχωριστά. 105 πρώτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Γίνεται δεκτή. 107. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα υπάρξει έλεγχος για την 107. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Πράγματι. Έγινε δεκτή. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 109. Τέλος. Γίνεται δεκτή η 109. 115. Κάτι είπε η κυρία Μακοβέη χωρίς μικρόφωνο, δεν την ακούμε. Δεν παραπονέθηκε κάποιος κυρία Μακοβέη. Τι ακριβώς είναι το πρόβλημα. Εξακολουθεί να μιλάει εκτό μικροφώνου η κυρία Μακοβέη. Κοιτάξτε, αν έχετε κάποιο πρόβλημα πρέπει να το λέτε αμέσως μετά την ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επανέλθουμε πίσω στην ψηφοφορία της τροπολογίας στην οποία αναφέρεστε. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 105. Άρχεται η ψηφοφορία. 105. Είναι πρόβλημα αυτό, λέει. Τέλος της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Τι να σας πω, εγώ ήμουν σίγουρος, λέει ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να μου το λέτε αμέσως. 115. Who is in favor? 150 υπέρ. Αποχές. Δεκτή. 116. Α, για μια στιγμή. Θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος για την 115. Συγγνώμη, 115 ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος της ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Uh, Κοιτάξτε, όταν uh, είναι 14 υπέρ και 12 κατά είναι δύσκολο λίγο για να είμαι σίγουρος και γι' αυτό έχουμε και τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Λοιπόν, 116 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 117 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 117. Uh, closed. Τέλος της ψηφοφορίας. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι δεκτή. <laughs> Okay. 118. 118. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 120. Ψηφίζουμε. Τέλος. Δεκτή. Η 121 καταπίπτει. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Η 122 καταπίπτει, η 123 καταπίπτει. Περνάμε τώρα στην 131. Όλες οι άλλες έχουν καταπέσει στην 22, 21 σελίδα μάλλον 131 υπέρ. κατά αποχές δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 134 Τέλος της ψηφοφορίας. 135 υπέρ. Κατά. Αποχής δεκτή. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 137 μέχρι 143 προτείνω να ψηφίσουμε ομαδών, σαν συμφωνείτε. Εντάξει, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 5, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Α, όχι, έχουν καταπέσει οι επόμενες. Περνάμε στην 146, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 147 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απερίφη. 148 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 148. Τέλος της ψηφοφορίας. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές δεκτή 157 υπέρ κατά αποχές δεκτή 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 159. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 164 καταπίτη Α, όχι, όχι, δεν έχει καταπέσει, οπότε ψηφίζουμε την 164. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 166. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 171. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 172. Υπέρ. Η 171 έγινε δεκτή θυμίζω, σαφώς. Τώρα, 172, επαναλαμβάνω υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 137, υπέρ. Συγγνώμη λέει 173 διορθώνει. Υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 175, υπέρ αποχές, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 177 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 178 υπέρ, κατά, αποχές, καταμέτρηση, έλεγχος, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 ε, μέχρι 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 185 υπέρ κατά 185 ψηφίζουμε ψηφίσαν όλοι πέρας ψηφίσουμε από κοινού 186 με 189, συμφωνείτε. Υπέρ, ποι είναι υπέρ, ποι κατά, αποχές, εγκρίνεται. 190, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 192, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομοδοτήσεις των Επιτρόπων. Ντεβε. 1 έως 8. Όλες μαζί, αν συμφωνείτε. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται απασχόληση. 1 έως 15 είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο. 1 έως 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μεταφορών 1 έως 14. Λίμπε. Ένα με τρία. Είναι υπέρ. Κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Πολιτιστική. Ένα έως πέντε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ένδυ. Ένα έως δέκα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΑΦΕΤ. Προηγούμενο 1. Υπέρ. Against. Abstention rejected. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 με 4. Υπέρ. Κατά εγκρίνονται. ΑΦΕΤ 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 6 καταπίπτει. 7 με 9. Όλες μαζί. Πίνε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος. Περιφερειακή. Ένα με τρία. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι 4, 5 υπέρ. Φωτά. Αποχές. Απορρίπτονται. Περιφρακή. 6 με 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γυναικών. 1 έως 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 1 έως 6. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ελίας. 1 έως 10. Όλες μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ολογικές παραγραφή. 194 υπέρ κατά Αποχέ, απορρίπτεται 195 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 196 υπέρ κατά απόχέ. εγκρίνεται 197 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά θα κάνουμε κατά μέτρηση 198 υπέρ ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρασε ψήφισαν όλοι πέρασε 199. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πέρασε. Εγκρίνεται μπορούμε να ψηφίσουμε από 200 203. Είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 204. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 205. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτονται. 206. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 206. Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτωτο. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 213 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 213 εγκρίνεται. 214 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Vote is closed. ψηφορίας. 25-2. Συγχαρητήρια. Herzlichen Okay. Ένα μικρό διάλειμμα. Now, number five. Περνάμε κατευθείαν στι ψηφορίε. Θα μπορούσαμε να τα ψηφίσουμε μαζί τι τροπολογίε 1 έω 6, αν συμφωνείτε. Αν συμφωνείτε. το σημείο 5. Ειδικέ εκθέσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο τη απαλλαγή τη Επιτροπή 2010. Μαζί οι τροπολογίε 1 έω 6 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνονται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα για το σύνολο του ψηφίσματο όπω τροποποιήθηκε. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Vote Uh, Και συνεχίζουμε με την απαλλαγή για το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη. Ο συνάδελφος Έρεν Χάουζερ είναι ο εισηγητή, δεν επιθυμεί να πάρει το λόγο. Και περάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ψηφοφορία λοιπόν. No. Um, citation 7. Amendment number Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Σύνδρο τη, τη, τη, το, την πρόταση. Ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορίας. As a whole, electronic vote is closed. Πέρας. Πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών. Ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία. Δεν ψηφίσατε όλοι ακόμα. Τώρα πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 17. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 17 παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας της Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Γιατί 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές να το ελέγξουμε γιατί την τροπολογία 21. Αν ψηφίσετε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 και 23. Α, όχι, 22, 22 εγκρίνεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. 23 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές, ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Έναρξη ψηφοφορίας, αν ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26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 ψηφοφορίας, μάλλον. Αν ψήφισατε όλοι, πέρας. Έγκρινεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατά πίτη 37. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε παρακαλώ. Για την 38 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 40 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές παρακαλώ. Με την 40 ηλεκτρονικό έλεγχο. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας τη ψηφοφορίας. 41. Η 40 εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ με την προφορική τροπολογία της κυρίας Μακοβέ. υπέρ κατά αποχές Να το ελέγξουμε παρακαλώ για την 44 ψηφίσατε όλοι πέρασε εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές ας το ελέγξουμε για την 45 παρακαλώ ηλεκτρονικά εννοώ αν ψηφίσετε όλοι πέρας της Δεν ήταν σαφές συγγνώμη 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 53 υπέρ. Η 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά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 Okay. 63 Ενδεχόμενη συμβιβαστική τροπολογία προφορική που καλύπτει αυτές τις τέσσερι ε, τροπολογίες. Σας την έχουμε μοιράσει. Διαδικαστικό εισηγητής. Θα ήθελα να πω ότι 63, 64 και 65 έχουν καταχωριστεί ως προφορικές τροπολογίες. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα, λοιπόν. Η προφορική τροπολογία την έχετε λάβει όλοι σα. Ωραία, τότε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία που περιλαμβάνει αυτέ τι τρεις ε, τροπολογίες υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να σηκώνετε καλά το χέρι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ. Όχι. 66, 66. Συγγνώμη, την ξέχασα. 66. Covering those four amendments. Which are these? Καλύπτει τις τέσσερις τροπολογίες αναφέρεται. Δεν γίνεται προφορική τροπολογία στην 66. Να ψηφίσουμε την 66. Για να είμαστε σίγουροι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε για την 71 παρακαλώ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αν ψήφισατε όλοι, πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 74 να το ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 74. Έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 77 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ο εισηγητής θέλει να πάρει το λόγο. Μία τεχνική διόρθωση. Δεν είναι 12% το ποσοστό, αλλά 14%. Μάλιστα με μία ε, διόρθωση. Σα ευχαριστώ. Στην 77 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπέρ 78. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 80. Υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε για την 80. Έναρξη ψηφοφορίας. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Α, περισσεύει ένας από το ΕΛΚ τώρα. Τώρα μάλιστα, είμαστε καλά. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Η 81 υπέρ. Υπέρ κατά. Δεν ήταν σαφές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 81 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 82 υπέρ. Για την 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ. Κατά αποχές Ας το ελέγξουμε για την 84 ηλεκτρονικά. Check is closed μέρας Εγκρίνεται. 85. πέρκατα κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ψηφίσουμε την 85 ηλεκτρονικά, να το ελέγξουμε. Την 85, ηλεκτρονικός έλεγχος, αν ψηφίσετε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 10 καταπίπτει η 11 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε για την 11 έναρξη ψηφοφορίας ψηφίσατε όλοι Rejected. Number 12 with oral amendment. Who is in favor? Abstention is taken. Number Αποστολές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. In block 15 to 8 if you like in block. Και τώρα 15 μέχρι 8 ε, όλες μαζί αν δεν έχετε αντίρρηση υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται. opinion, one in favor. Υπέρ, κατά, μετά, αποχές και απορρίπτεται. Δεύε, μόνο δύο. Όλες μαζί, εάν ε, θέλετε να ελέγξουμε για το υπαριθμόν 1 αν και είναι, γίνεται, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, έλεγχος, έλεγχος λέγω, έλεγχος. Uh, they were not participating, the colleagues. Sorry for that. It is... Συνάδελφοι, ψηφίσατε διότι εγκρίνεται. Οπότε, οι υπόλοιπες θα γίνουν όλες μαζί. 2 με 11. Ποιοι είναι υπέρ. Τώρα, όχι. 2 με 10. 2 έως 10. Ποιοι είναι υπέρ. 2 έως 9 λέει τώρα ο Πρόεδρος. Όλες μαζί. 2 έως 9. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Και εγκρίνεται. 10 τώρα. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 10. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται. Η, της ΔΕΒΕ υπερχμών 11, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε. Όσον αφορά την πρόταση ψηφίσματος συνολικά, όπως τροποποιήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ψηφίζουμε τώρα. Vote is closed. Και ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Äh, Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εισηγητή, ο Στόλικο Λιμπράτσκι, θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Λιμπράτσκι. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem w zasadzie bardziej zabrać głos ze Ήθελα το λόγο γιατί θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για μια εξαιρετική μορφή συνεργασίας και τις Γενικές Διευθύνσεις και της Κομισιόν εννοώ και τη Γενική Γραμματεία του Κοινοβουλίου μας πάντα διέθεσαν πληροφορίες, χρόνο, επικοινωνία, ήταν διαθέσιμοι όλοι. Να ευχαριστήσω τους κυρίους κυρίους Μπλέσα και Κούρχαρτ γιατί η δική τους συνεισφορά ήταν καθοριστική. Äh, Ευχαριστούμε τον εισηγητή και μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Δεν θα ψηφιστεί γιατί δεν είναι νομότυπη και το περνάμε λοιπόν στην συνολική ε, ψηφοφορία για το σύνολο της ε, απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε λοιπόν. Έναξη ψηφοφορίας. Αν ψήφισατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας. Okay. I continue in English. 4 to 8 could be in a block vote if you accept. No? 4 to 7. 4 με 7. Όχι από κοινού, όχι ξεχωριστά. Η 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Για την 4 μόνο ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Α, ηλεκτρονικός έλεγχο για την 9. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Και 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Έλεγχος ηλεκτρονικός 13 και 16 μαζί. Ψηφίζεται. Τελειώσατε. Τέλος. Δεκτές. Δεκαεφτά υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεκαοκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεκαεννέα υπέρ κατά, αποχές, δεκτή. 20. Το πρώτο τμήμα δεν γίνεται αποδεκτό, το δεύτερο τμήμα το ψηφίζουμε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20. Όλη η τροπολογία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 Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, παρακαλώ. Jeder abgestimmt, dann ist die Abstimmung geschlossen. Αν ψηφίσατε όλοι, ολοκληρώνεται η ψηφοφορία και εγκρίνεται. Με 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Εντάξει. Για την 30. Ηλεκτρονικός check is check is... Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Να επαναλάβω. Γιατί 33. Υπέρ. Υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Άποχες. Να το ελέγξουμε για την 33 ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Για την 35. Α, συγγνώμη, την 34. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ Γιατί 35 παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται ωραία και τώρα περνάμε σε ξεχωριστή ψηφοφορία από το ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 36 τότε. Όχι. Η 36, 38, η 37, 39 κατά πίπτων. Και συνεχίζουμε με τη 40. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ ηλεκτρονικά να το ελέγξουμε. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Όταν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται η 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι και βεβαίω. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, έλεγχος. Ψηφίστε. Πέρας. Σαφέ το αποτέλεσμα. Η 42. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 44. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 45. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε κιόλας. Για την 45. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Αυτό για τη 45. 29. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46. Α, καταπίπτων.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 Αν ψηφίσατε όλες σας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχο. Πολύ ωραία. Έλεγχο. Για την 57. Αν ψηφίσατε όλοι, yes. Εγκρίνεται. Με οριακό αποτέλεσμα. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ για την 59. Πέρας της φιβουρίας. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 64. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτοντα. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 70. Ξεχωριστά. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ας το ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Έναρξη ψηφοφορία. Αν ψήφισατε όλοι, πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται, αλλά αυτό ελέγξουμε. Για την 79. Την 71, συγγνώμη. Έναρξη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Αν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. 72 υπέρ. Κατά. Αποχέ 70 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ για την 74 πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ. Κατά. Αποχέ, Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. απόχέ. Να το ελέγξουμε για την 78 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86. Α, 85, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Παρακαλώ να το ελέγξουμε. Την 86 ηλεκτρονικά την ψηφίζουμε. Αν ψηφίσατε όλοι για την 86. Εγκρίνεται. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε για την 88. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οι 92 και 90 καταπίπτουν. 94 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ για την 95 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της, της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με διαφορά. 97 υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη. Έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Το ζήτησε η κυρία Γκρέσλε για την 97 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. σημειώνεται ότι το πρώτο τμήμα μέχρι το prize. Αν έχετε κάποια ένσταση θα πρέπει να ψηφίσουμε στο σύνολο της τροπολογίας. Δεν το αποτέχεστε. Ωραία. Θα ψηφίσουμε όλο το 97. Κυρία Κρέσλε. Υπάρχει μία έκθεση για το ταξίδι αυτό, άρα επί του προηγουμένου είναι λάθος αυτή η πρόταση. Άρα είναι λάθος αυτό που αναφέρεται ότι δεν έχει αναφερθεί ε, στο Κοινοβούλιο ποιο ήταν ο σκοπός και το όφελος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ζήτησα να αναφερθεί αυτή η τελευταία μισή πρόταση. Το πρόβλημα λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, είναι ότι δεν υπάρχει σαφήνεια στην συνάδελφε Γκάιερ. Στα γερμανικά ήταν λίγο πιο σαφέ. Εντάξει, κοιτάξτε, καταψηφίζουμε και τα δύο, άρα είναι απλά τα πράγματα. Σε τμήματα ψηφοφορία. Για το πρώτο και για το δεύτερο τμήμα. Για το πρώτο τμήμα λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε λοιπόν για το πρώτο τμήμα. Hat jeder abgestimmt? Ψηφίσατε όλοι. Πέρα λοιπόν τη ψηφοφορία. Με ισοψηφία λοιπόν απορρίπτεται η τροπολογία. Για το δεύτερο τμήμα λοιπόν δεν υπάρχει, δεν γίνεται ψηφοφορία. Ωραία, και τώρα περνάμε στην 98, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρας της υποφορίας. εγκρίνεται για την 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 102 ηλεκτρονικά ψηφίζουμε αν ψηφίσατε όλοι ολοκληρώνεται η ψηφοφορία για την 102 εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 103 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 106 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 107. Ηλεκτρονικός έλεγχος ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Για την 113 παρακαλώ. αν ψηφίσετε όλοι. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Απορρίπτεται. Από 14 στα τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να το ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Εγκρίνεται με διαφορά. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές και την 115 παρακαλώ να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελεκτρονικό check is geschlossen. Πέρας. Εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για 117. Αλλά να σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. Έλεγχος ηλεκτρονικά. Αν ψηφίσατε όλοι, να ολοκληρώσουμε τον έλεγχο. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. 121 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 122. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 124. Πέρας. Εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές και αυτό δεν είναι σαφές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 126. Ψήφισατε όλοι. Για την 125, συγγνώμη, για την 125. Εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό είναι οριακό. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ για την 126. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Αυτά για την 126. 127 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται 131 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικά για την 131 πέρας εγκρίνεται 132 υπέρ Απορρίπτεται. 133. Υπέρ, κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε, θα το ελέγξουμε για την 135 έναξη του ελέγχου της ειρηνικής ψηφορίας. Αν ψηφίσετε όλοι, Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εκατόν τριάντα έξι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εκατόν τριάντα επτά. Υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε. Για την 135. Είναι 137, συγγνώμη. Ηλεκτρονικός έλεγχο. Πέρασε. Εγκρίνεται. 138. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 139, πρώτο τμήμα. Υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικό έλεγχος αν θέλετε. Για τον 141. πέρα. Εγκρίνεται. 142. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Mm, δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος, αν θέλετε, για την 142. Πέρας τη ψηφοφορία Εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 148 παρακαλώ. Έναξη ψηφοφορία. Αν ψήφισατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Πάμε για την 149 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισατε όλοι. Ναι, είναι σαφής, ε, σαφές το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται. Ποιος κουράστηκε, δεν είμαι σίγουρος. Αν θα σηκώνατε όλοι τα χέρια σας, θα ήταν πιο σαφή τα πράγματα. 150. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 151. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. το ελέγξουμε ηλεκτρονικά αν θέλετε για την 154. Αν ψηφίσατε όλοι. Ναι, ήταν ωριακό το αποτέλεσμα, από ό,τι βλέπετε. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Mm. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 155 υπέρ. Κατά. 155 υπέρ. Κατά. Mm. Αποχές εγκρίνεται. 156 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157. Προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 160 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Ας το ελέγξουμε για το πρώτο τμήμα της 160 παρακαλώ ποινική ψηφοφορία Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε και το δεύτερο τμήμα. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Όπως σας είχα πει. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Για την 161 παρακαλώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Α, ήταν μάλλον σαφές το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 164 ηλεκτρονικά παρακαλώ εγκρίνεται Εκατόν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 166 παρακαλώ πέρας εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 170 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα η συνολική ψηφοφορία όπως τροποποιήθηκε το κείμενο ηλεκτρονικά παρακαλώ έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αν ψηφίσατε όλοι ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Αν έχετε κι άλλη ενέργεια, να συγχαρούμε τον εισηγητή. Και περνάμε στο τελευταίο σημείο. Vote. Έγκριση τέλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ε, πειθαρχημένη αυτή η εργασία και τα λέμε αύριο. Εκτός και αν θέλετε κάτι να παρατηρήσετε, μάλιστα, διακοπή λοιπόν της συνεδρίασης, τα λέμε αύριο το πρωί στις 9. Okay.